Και βεβαίως ο στόχος είναι να επιτύχουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά η οποία θα είναι φιλική προς το χρήστη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Αυτό σήμανε και το τέλος της συζήτησής μας. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο από τις 9 μέχρι τις 2 και το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνατε μέχρι τόσο αργά. Ευχαριστή και τους διερμηνείς ο πρόεδρος και αυτό σημαίνει και το τέλος της συνεδρίασης.